Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Η πρώτη ψηφοφορία αφορά καταπήγον ψήφισμα έξι ομάδων για την Ρουάντα, για την περίπτωση της ε, Ιγκαμπίρα. Ψήφισμα, λοιπόν, συνολικά ψηφίζουμε υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Επόμενο ψήφισμα για το Σουδάν. Ψήφισμα επτά ομάδων ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο της ε, παραγράφου 6, αλλά έχουμε προφορική τροποποίηση από τον κύριο Σβόμποντα, ο οποίος και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, προτείνω να τροποποιήσουμε την παραγράφο 6 του ψηφίσματος, οπότε στο τέλος της παραγράφου να, προτείνουμε, να προσθέσουμε την φράση και ιδιαίτερα ανησυχητικό και ύστερα να προσθέσουμε τέσσερα ονόματα όπως αναφέρεται στον κατάλογο ψηφοφορίας.